Right, Αγαπητοί συνάδελφοι, μήπως θα μπορούσα να ζητήσω από όλα τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ και ΛΥΜΠΕ και λοιπόν persons to eventually leave our committee room. Να αποχωρήσουν από τη αίθουσα της Επιτροπής μας ησύχως. Επίσης μπορείτε να μιλάτε και λιγότερο την ώρα που αποχωρείτε. So, we're running slightly late, so let's continue. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Συνεχίζουμε λοιπόν σημείο 5 στην ημερησία διάταξη. Ε, πρώτη συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Νόριτσα Νίκολαη. Ε, παρευρίσκεται μάλιστα συστάσει προ το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΕΔ σχετικά με τι διαπραγματεύσει για τη Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αζερβαϊτζάν ήθιστε στην Επιτροπή μας να λέμε τι περιμένουμε από τους διαπραγματευτές έτσι ώστε να ε, διατηρηθεί η διαδικασία ε, ε, που παγίως τηρείται. Μπορείτε να θυμάστε ότι το διαβριμένο Προεδρείο ε, ανέβαλε κατά δύο μήνες το χρονοδιάγραμμα για να ε, ακούσουμε τα αποτελέσματα της αντιπροσωπείας που θα μεταβεί στο Μπακού το Μάιο ε, και σχετικά με την απελευθέρωση κάποιου κρατουμένων. Τελικά το Συμβούλιο έστειλε έγγραφα για τις διαπραγματεύσεις αυτές επιτέλους και είναι έγγραφα στα οποία εμείς δικαιούμαστε να έχουμε λόγω και συμμετοχή και στο μέλλον θα πρέπει να αποφεύγονται τις δυσκολίε, λέει το διευρυμένο Προεδρείο. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Νικόλαη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια νέα συμφωνία είναι αυτή. Πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι σχέσεις μας με το Αζερβαϊτζάν διέπονται από μια συμφωνία του 1999 και έχει περάσει τόσους χρόνους. Είναι από τους βασικούς εταίρους, εμπορικούς εταίρους, σας θυμίζω, το Αζερβαϊτζάν. Πάνω από 50% του συνολικού εμπορίου του Αζερβαϊτζάν γίνονται με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 55% ε, είναι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα αυτή, επί του συνόλου των εξαγωγών. Άρα το εμπόριο κυριαρχεί και οι οικονομικές μας σχέσεις είναι αρκετά ισχυρές πέρα από τις πολιτικές και γενικότερες. Όπως σας είπα, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ε, διέπονται από μια συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας που ανάγεται στο 1999. Η συμφωνία αυτή είναι μη προτιμησιακή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποιες ευνοϊκές ε, ρυθμίσεις. Ε, υπάρχουν και ποσοστώσεις στο διμερές εμπόριο. Πέρυσι άρχισε η διαπραγμάτευση, η οποία συνεχίζεται. Και ελπίζω οι συστάσεις μας να ληφθούν υπόψη και να είναι σημαντικές στην έκθεσή μου γίνεται λόγος για την επίλυση και την έρευση που είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Ε, οι βασικές αξίες για μας παραμένουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία φυσικά και όλες οι αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας η προώθηση και τη συνειδητοποίηση μεταξύ ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αζέρων ε, ως προς τις νέες πολιτικές, νέες, τις, ε, νέες ευκαιρίες κλπ. Επίσης, σύμφωνα με την πολιτική μας δήλωση και την παράδοσή μας, εμείς υποστηρίζουμε την εδαφική ακαιρεότητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα. Και σύμφωνα με την ομάδα του Μίνσκ ε, και οι δύο πλευρές και σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες και τα ψηφίσματα ελπίζουμε να έχουμε σύντομα μια ειρηνική διευθέτηση της σύραξης στην περιοχή. Uh, Για μας τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν βασική ανησυχία και μέλημα. Πρέπει να ενισχύσουμε το ισχύον πλαίσιο ε, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και θέλω να καλωσορίσω το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο και την υποστήριξη που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Όπου περιμένουμε να έχουμε δικαιοσύνη για όλους και ειδικέ διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της ε, φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ε, επίσης εμείς ε, εκτιμούμε πάρα πολύ και προάγουμε την πολυφωνία ε, στον τύπο και στα μέσα ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές ε, του Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να βελτιωθεί ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στην κοινωνική ζωή. στα επιχειρηματικά και εμπορικά σχέδια θα υποστηρίξουμε το Αζερβαϊτζάν να κάνουν ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της αγωνιστικότητας, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη διαφοροποίηση της οικονομίας. Υπάρχει ανάγκη ε, να ενθαρρυνθεί επιχειρηματικότητα και ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα ε, επέλθει ανάπτυξη μέσω Φυσικά η ενεργειακή συνεργασία κυριαρχεί στη συμφωνία. Αυτή τη στιγμή το Αζερβαϊτζάν για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς, σημαντικούς και στρατηγικούς εταίρους. 5% περίπου το πετρελαίο εισάγουμε από το Αζερβαϊτζάν και διαδραματίζει και ρόλο κλειδί στη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου από την Κασπία από τους νότιους ε, αγωγούς φυσικού αερίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποστηριχθεί αυτή η πολιτική με συνεργασία και στα ενεργειακά, διότι αυτό δεν είναι μόνο προς όφελος της οικονομίας και των δύο πλευρών, αλλά είναι και μια ευκαιρία εξασφάλιση του ανεφοδιασμού και της ασφάλειας γενικά στην περιοχή. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω και τον ε, αγωγό Trans Anatolian. Είναι ένα διεθνές έργο ε, εκεί που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν ε, διαμέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, να τονίσω δύο πράγματα που θεωρώ πολύ σπουδαία. Για να στεφτεί με επιτυχία αυτή η συμφωνία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να αυξηθεί η κοινοβουλευτική συνεργασία. Το τονίζω αυτό. Το τελευταίο διάστημα συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τους ομολόγους μας από την Αζερική Βουλή και ελπίζω να εδραιωθεί και μια αναβαθμισμένη κοινοβουλευτική δομή συνεργασίας για να υποστηρίξουμε έτσι την πολιτική, την οικονομική συμφωνία αλλά και τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Ελπίζω κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να συνεργαστούμε καλά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να συνεχιστεί αυτή η αγαστή συνεργασία που είχαμε. Και η κατάσταση ελπίζουμε να βελτιωθεί στο Αζερβαϊτζάν, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται κοινή προσπάθεια, συνεργασία, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερβαϊτζάν. Αυτή τώρα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Περιμένω τις τροπολογίες σας και ελπίζω να έχω την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων για να προχωρήσουμε σε σαφείς συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή με το Ζερβαϊτζάν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Νικολάη. Και τώρα το λόγο θα πάρουν οι σκιώδεις και οι υπόλοιποι που θέλουν. Κάποιον ξέχασα. Α, τι έγινε το μεταξύ. Μάλιστα. Γκόμες. Δύο με τρία λεπτά έκαστος. Κάτι πήρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξ ε, του ε, των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Φάμπι Λόπες, Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάη για το σχέδιο έκθεση. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να εστιάσω στο κεντρικό θέμα που αναφέρατε και εσά και εσεί, δημοκρατία, κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, Στι διαπραγματεύσει μας με το Αζερβαϊτζάν. Για μας, τους σοσιαλιστέ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν θα υπάρξει έγκριση χωρίς σαφή απτή και αποδεικνυόμενη απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Είναι το μήνυμο για τους σοσιαλιστές για να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε στις αρχές του Αζερβαϊτζάν παλαιότερες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζουν την πλήρη συμβασμό των διεθνών ε, δεσμεύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιρροή ε, των θέσεων ε, στο την πλήρη εφαρμογή των, των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι οι υπερχόμενες προεδρικές εκλογές. Βλέπουμε ότι ε, δεν ακολουθούνται οι κατευθυντήριες νέες γραμμές και κάποιοι βασικοί υποψήφοι όπως ο Γιούγκα Μαμόντοφ είναι ακόμα στην φυλακή. Δεν υπάρχει ισοτιμία, δεν υπάρχει ελευθερία του. Συνέρχεστε ε, και ε, γι' αυτό ε, θα πρέπει και οι ελεύθερες και δικές εκλογές να είναι, ε, να είναι μοχλός για την έγκριση αυτής της έκθεσης. Κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ένα ειδικό μηχανισμό ακύρωση σε σχέση με τα, η αναστολή μάλλον, σε σχέση με τι θεμελιώδει ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στη Νέα Συμφωνία και ένα τελικό στοιχείο που επίση ε, θύχθη από τον εισηγητή, για την, ε, ε, από την εισηγήτρια για τη σύγκρουση Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ναι, βεβαίω θέλουμε να γίνει σεβαστή η ακυρεότητα και η κυριαρχία του Αζερβαϊτζάν, και το καθεστώ του Ναγκόρνο Καραμπάχ αμφισβητείται, δεν υπάρχουν για τα τις γύρω περιοχές που εξακολουθούν να κατέχονται από τις αρμενικές ε, δυνάμεις. Επίσης, είναι σαφές από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι αυτό πρέπει να επιστραφούν στο Αζερμπαϊτζάν. Όσον αφορά το Αζερμπαϊτζάν και την Ρωμανία, θα πρέπει να πούμε ότι δίνεται προτεραιότητα στο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και επίσης ότι στηρίζουμε την ομάδα ΜΕΝΣΚ της ΟΑΣΕ. Για μας λοιπόν η όρη αυτή είναι πολύ σημαντικό τμήμα της έκθεσης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κάτι πήρη. Και τώρα εξ ονόματος της κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάη για την ε, για τις προτάσεις της, ε, της πλήρης ε, και τα ευρήματά της. Το Αζερμπαϊτζάν είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε γεωπολιτικό επίπεδο. Ε, σε ζητήματα ασφάλειας της περιοχής και θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που δεν αναφέρθηκε στις συζητήσεις μας νωρίτερα ο ρόλος της χώρας αυτής ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με ε, τον ελεύθερο κόσμο, τις, τους διεθνείς θεσμούς ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η χώρα αυτή ε, πραγματικά ακολουθεί τις δυτικές αξίες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως ε, όταν είχαμε αποφασίσει να αναβάλουμε ε, την συζήτηση για τις συστάσεις ε, ε, περιμέναμε βεβαίως να γίνουν κάποια πράγματα ε, αμνηστία από τους πολιτικούς προκρατούμενους παραδείγματος χάρη με την ευκαιρία των 100 ετών των του εορτασμού για των 100 ετών για την ύπαρξη του, χώρα του Αζερμπαϊτζάν, ε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Στόλτς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ τον εισηγητή ο Σόλτς ε, Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα βεβαίω ε, ότι υπάρχει έντονη διασύνδεση με το τι συμβαίνει σε άλλε χώρε τη περιοχή, Αρμενία και Γεωργία. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι βεβαίω ε, και είναι προφανέ ότι το Αζερβαϊτζάν, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εταίρο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που γίνεται ε, για τη δική του οικονομική ανάπτυξη. Βεβαίως είναι κάτι που συνδέεται και με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και πρέπει να πω ότι είναι σαφές ότι οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας για τις περαιτέρω εξελίξεις ε, στις νομοθετικές διαδικασίες στη χώρα το, θα πρέπει οι συνταγματικές ε, μεταρρυθμίσεις να μεταφραστούν και σε συγκεκριμένη νομοθεσία ε, έτσι ώστε να πληρώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ECHR είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις της ΕΣΤΑ Είναι περίπλοκο περίπλοκη κατάσταση εκεί, στι διμερεί σχέσει που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε ε, τη συγκεκριμένη πραγματικότητα στη χώρα αυτή, σε κοινωνικό επίπεδο, να δούμε τι έχει επιτευχθεί και να επιφυλασσόμεθα για τις ε, μελλοντικέ εξελίξεις ε, στην σχέση αυτή. Βεβαίως συμφωνώ ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για μας, για τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Ευχαριστώ τον Χέλμουτ Σόλτς τον σκιώδη συγητή από η σκιώδη γίνει ένα ζώφκο από το ΕΛΚ μου ζήτησε να πω δύο λόγια στο όνομά τη. Η κυρία Σόφκο αυτή τη στιγμή είναι σε αποστολή στο Νεπάλ και ζητεί συγγνώμη που δεν μπορεί να παραστεί εδώ σήμερα. Αναγνωρίζει τη σημασία της μελλοντική ε, συνολικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερμπαϊτζάν η οποία θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο ε, για τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος, ενέργεια, ε, επενδύσεις. Ε, υπάρχουν διάφορα σχέδια για αγωγούς αερίου, ε, διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Ε, βεβαίως πρέπει να υπάρξει η σφαιρική συμφωνία, πρέπει όμως να εφαρμοστούν και οι βασικές αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου που πολύ σωστά αναφέρονται στην έκθεση. Επιπλέον Υπάρχει και ένα πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να δοθεί έμφαση κυρίω στην προσέγγιση συνεργασία με το Ροσμπατζάν, σα αφορά την ανθρωπίνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Αυτά είπε η κυρία Νισόφκο. Και τώρα η κυρία Γκόμε έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και μετά να μην το να εξετάζουμε τι επιμέρους περιπτώσει, τι συγκεκριμένε περιπτώσει. Ε, οι οποίες ε, ε, πραγματικά ε, αμφισβητούν άμεσα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κάτι Πύρη αναφέρθηκε στην απόφαση του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να απελευθερωθεί ο, ο κύριος Μαμαντάφ, ο οποίος είναι στη φυλακή επειδή είχε κριτικάρει την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου και έχει προσφύγει κατά της απόφασης και η ίδια προσφυγή δεν έγινε αποδεκτή από το δικαστήριο. Ξέρουμε ότι οποιαδήποτε κριτική όχι μόνο από πολιτικού, αλλά από δημοσιογράφου, οποιονδήποτε, οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσει το οτιδήποτε, ε, αντιμετωπίζεται με βία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην κάνουμε τίποτα όταν υπάρχει παραβίαση ε, καταφανή από χώρα όπω το Ζερβαϊτζάν, που είναι υπεύθυνη και για τη διαφθορά όπως πολύ σωστά είπε κύριε Νικολάη, όχι μόνο διαφθορά στο Αζερμπαϊτζάν, χρήματα δηλαδή που θα πρέπει να πάει στο λαό του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίπτωση της Μάλτας, ε, την οποία μπορέσαμε να ανακαλύψουμε στην ε, αποστολή μας στη Μάλτα. Υπάρχει μια τράπεζα που λέγεται Pilates Bank, που ουσιαστικά ξεπλένει χρήματα από το Αζερμπαϊτζάν της κυρίας Αλίεβα, του, του Υπουργού Εσωτερικών, δεν είναι μόνο διαφθορά στο Αζερβαϊτζάν, είναι και διαφθορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να μας απασχολεί αυτό. Αποφασίστηκε να, δοθούν, να δοθεί ένα δισεκατομμύριο ε, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, για έναν αγωγό από το Αζερβαϊτζάν στην Ιταλία. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, που έστειλαν επιστολές στην πακέτα Τράπεζα Επενδύσεων, αυτό θα δημιουργήσει χάος ε, σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για άλλη μια φορά. Ε, είναι πραγματικά παράδεκτο το γεγονός ότι ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εμείς δηλαδή, ξακολουθούμε να παραβλέπουμε τόσο σημαντικά στήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπε και η Κάτι Πύρη, θα πρέπει να το δούμε αυτό με βάση και το τι θα συμβεί στις εκλογές. Αν θα υπάρξουν δηλαδή οι ε, ίσες ευκαιρίες. Διότι ε, ακόμα και βουλευτές αυτού του κοινοβουλίου υπέστησαν, κυρώ, υπέστησαν επιπτώσεις από το, την κυβέρνηση του Ζερμπατζάν. Δεν μπορούμε πλέον να εθελοτυφλούμε. Ευχαριστώ. Κύριο Στέτινα για το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα μιλήσω ε, τσεχικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Θέλω να πω τα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της έκθεσης, και το δεύτερο για το Ορνό Καραμπάχ. Κύριε Εισηγήτρια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για τη λεπτομερή σας αναφορά σε αυτό. Θα μπορούσε να διατυπωθεί και πιο έντονα στην έκθεση αυτό το θέμα. Αναφέρεται κάποιους δημοσιογράφους, αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κυρώσεις ε, απέναντι σε ηθήνοντες ε, που έχουν κλείσει κάποια μέσα ενημέρωσης, το Radio Free Europe ή άλλες ε, εφημερίδες επιγραμμικές και το κανάλι TV Maidan. Γίνονται τρομερά πράγματα στο Αζερβαϊτζάν. Αυξήθηκε ε, σε πενταετή φυλάκιση η ποινή ε, για το αδίκημα της εξύβρισης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Όπου βρίσκει κανείς ποινικού κώδικες με τέτοιες διατάξεις, το καθεστώς είναι δικτατορία. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Αυτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τον Αγκόρνο Καραμπάχ δεν έχω χρόνο να μιλήσω από ό,τι βλέπω. Ε. Ευχαριστώ κύριε Στέτινα. Η κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη, γιατί η συγκητρία είναι από τη δική μου πολιτική ομάδα. Απλώς να πω ότι ε, ε, ό,τι και να πούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι λίγο. Ο κύριος Στέτινα, μήπως να κλείνετε το μικρόφωνο σας, λέει ο πρόεδρος. Thank you. Ωραία. Επήλθε και πάλι η σαφήνεια στο σύστημα και φαίνομαι και στην οθόνη. Δεν θα επιμείνω, ούτε έχω να προσθέσω πολλά όσα είπε η κυρία Νικολάη, αλλά ε, όσο και να τονίζουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν φτάνει ε, όταν συζητούμε για το Αζερβαϊτζάν. Θα μπορούσαμε λίγο να διευκρινίσουμε ε, ποιους όρους βάζουμε ε, για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Λέει το κείμενο ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ε, τι θα πει αυτό, είναι επαρκή τα βήματα αυτά και πώς μπορούμε να πιέσουμε πολιτικά και με άλλους τρόπους και να βαρύνουμε έτσι ώστε όλοι οι ε, πολιτικοί κρατούμενοι που κρατούνται αδίκως να φερθούν ελεύθεροι. Επίσης, να ε, βάλουμε και κάποιους όρους για την κοινοβουλευτική συνεργασία. Βεβαίως και μπορεί να γίνει ευκαιρία αυτό, αλλά μόνο εφόσον οι εκλογές είναι δίκαιες και οδηγούν στην ευάθυνση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι σε αυτή τη χώρα η πρώτη κυρία είναι και αντιπρόεδρος της δημοκρατίας. Okay. Thank you, Ευχαριστώ, Μαρίτσι. Τελειώσαμε αυτό το σημείο. Mr. Devine, is there from the... Oh, there you are. Από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ξέχασα τον κύριο Ντεβίγε. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση να σα ενημερώσω για την κατάσταση πρόοδου των διαπραγματεύσεων μα για την νέα διμερή συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν. Και σα ευχαριστώ, κύριε Νικολάη, για το σχέδιο σύστασης. Δύο ε, λόγια για το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Έπρεπε να ανανεωθεί η 20 ετής αυτή η συμφωνία που έχουμε με αυτή τη χώρα. Βέβαια πολλά πράγματα έχουν συμβεί στην 20 ετία αυτή και οι σχέσεις μας έχουν εξελιχθεί. Ιδιαίτερα η ανατολική εταιρική σχέση, ε, της οποίας αποτελεί τμήμα το Αζερβαϊτζάν. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία, όπως η διευκόλυνση θεωρήσεων και η συμφωνία ε, ε που έχει συμφωνηθεί από το 2014, καθώς και το πρόγραμμα συμμετοχής του Αζερβαϊτζάν στα προγράμματα της Ένωσης και στους οργανισμούς ε, μέσα στο πλαίσιο μιας εταιρική σχέσης κιν, κινητικότητας. Βεβαίως, το, οικονομικά το Αζερβαϊτζάν είναι στρατηγικός εταίρος της Ένωσης και η κλειδί για τον διάδρομο φυσικού αερίου ε, που όπως ξέρετε είναι κλειδί για τη διαφοροποίηση. Αυτός ο διάδρομος έχει, θεωρηθεί, έχει μάλλον οριστεί ως ε, προτεραιότητα κλειδί από το ίδιο το Συμβούλιο από το 2015. Είναι βέβαια σταθερός τέρος σε δύσκολη σε περιοχή όπως τα προς τα βορρά έχει τα σύνορα με το Τεγκιστάν. Έχουμε βέβαια την, και την ε, Συμφωνία για Στρατηγική Εταιρική Σχέση και ξεκινήσαμε τη διαπραγματεύση ε, στις αρχές του 2017. Είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία θα ενταχθεί στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ε, πολιτικής ανατολικής γειτονίας και αυτό που θέλουμε είναι να αναπτυχθούν νέες ευκαιρίες με το Αζερβαϊτζάν για ε, ε, εμπλοκή σε διάφορους τομείς όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, η παιδεία αλλά και επίσης σε τομείς όπως τα κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και ευρύτερα στο οικονομικό πεδίο. Δύο σημαντικά ε, γεγονότα έγιναν. 24 Νοεμβρίου επιτυχής ε, διάσκεψη κορυφής ε, με την Ανατολική Εταιρική Σχέση με συμμετοχή του Πρόεδρου Αλίεφ και το Συμβούλιο Συνεργασίας στο οποίο προείδρευσε η κυρία Μογκερίνη και ο Υπουργός Εξωτερικών Αγιορφέκτοτε. Είχαμε διάφορες διαπραγματεύσεις Είχαμε 7 γύρους από τη δική μας πλευρά και 2 γύρους ε, διαπραγματεύσεων στην πλευρά του εταίρου. Ε, σύντομα, ε, να πω ότι έχουμε σημαντική πρόοδο, ότι... Η συμφωνία θα περιλαμβάνει διατάξεις για το πολιτικό διάλογο και την ασφάλεια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να τονίσω πως υπάρχει και ένα στάνταρ τίτλος πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ας πούμε για τα πρόσφατα θέματα εσωτερικών. Δυσκολίες ε, παραμένουν ε, στο Διεθνές Δικαστήριο και σε άλλα ε, θέματα. Τομεακά όμως, το τελευταίο των έξι γύρων έγινε την περασμένη Παρασκευή και εννέα κεφάλαια έχουν ε, για την ώρα ολοκληρωθεί. Περιβάλλον, επιστήμες, ε, προστασία καταναλωτή, απασχόληση, κοινωνική πολιτική, ε, βιομηχανική πολιτική, νεότητα, τουρισμός, αθλητισμός και παιδεία. Και σχεδόν κοντεύουμε σε συμφωνία για το θέμα του πολιτισμού, της πολιτικής πολυμορφίας και του διαπολιτιστικού διαλόγου, στις μεταφορές και στην ενέργεια. Τέλος, ε, και για το τμήμα του εμπορίου είμαστε, έχουμε κάνει δύο γυρούς διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή Ίντα ενημερώθηκε από τους συναδέλφους της Κομισιόν τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμής είχαμε συζητήσεις για την εμπορία αγαθών, βιομηχανικά πρότυπα, διαφάνεια, ε, πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, φυτογενομικά, ε, ε, τελωνία, επίλυση διαφορών, ανταγωνισμός, δημόσιες προμήθειες, βιώσιμη ανάπτυξη και αμοιβαία διοικητική αρρωγή σε θέματα τελωνιακά. Είχαμε καλή ε, συνεννόηση το τελευταίο γύρο. Μία συμφωνία έγινε για τα τελωνιακά θέματα, μηδέα αρρωγή για τα θέματα των τελωνίων, αλλά είναι σαφές ότι η μη συμμετοχή στον ΠΟΕ του Αζερβαϊτζάν δημιουργεί δυσκολίες και είναι βέβαια πολύ σημαντικό για το Αζερβαϊτζάν να θέλει να αναπτύξει αυτό που προτίθεται να κάνει, δηλαδή να είναι ένας κόμβος στον για τους εμπορικούς διαδρόμους με την Ανατολή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νικολάη, να κλείσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Βεβαίως, ελπίζω πως όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ε, συνεννοηθούμε είναι να συνεργαστούμε και πραγματικά ε, καλωσορίζω αυτή τη συμφωνία που είναι τώρα ε, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής καλής γειτονίας και καλωσορίζουμε το Αζερβαϊτζάν σε αυτήν την πολιτική καλής γειτονίας. Για μας είναι μια δυνατότητα να αξιολογήσουμε πιο ανοιχτή προσέγγιση από τις ε, αρχές του Αζερβαϊτζάν στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον επόμενο μήνα που θα είμαι στον Πακού θα είμαστε όλοι η αντιπροσωπεία μας και θα συζητήσουμε με τους ε, εκπροσώπους του Αζερβαϊτζάν. Ελπίζω πως σύντομα θα συμφωνήσουμε για την απελευθέρωση κάποιων πολιτικών κρατούμενων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Φωτίγκα που τονίζει το θέμα τα ασφαλείας στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως ε, γνωρίζω το Αζερβαϊτζάν αποτελεί χώρα διέλευσης για Ε, για τη στρατολόγηση ανθρώπων που συμμετέχουν στο πόλεμο της Συρίας και από πλευράς του ε, Ασάτ και από πλευράς του Ίσης. Θα ελέγξουμε λοιπόν τι συμβαίνει εκεί. Περιμένουμε λοιπόν τις τροπολογίες και ελπίζω πως θα μπορέσουμε πράγματι να βελτιώσουμε τη σχέση μας γιατί είμαι βεβαία πως αυτό θα είναι προς όφελος όλων ειδικά σε ένα τόσο τεραγμένο κόσμο, σε μια τόσο τεραγμένη περίοδο και με μια ισχυρή ε, Ρωσία, όπως έδειξαν οι Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να έχουμε καλή συνεργασία με το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, 4 Απριλίου λίγη προθεσμία ε, για τις τροπολογίες. Πάμε στα δύο επόμενα θέματα, 6 και 7, από κοινού. Σύναψη συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αφενός και της Αυστραλίας αφετέρου. Τον Αύγουστο του 2017 υπεγράφει η συμφωνία αυτή. Έχω μάθει ότι κατατέθηκαν 62 τροπολογίες, 22 Φεβρουαρίου έληξε η ε, προθεσμία. Ο Φρανσίσκο Μίγιαν Μον είναι εισηγητής, έχει προτείνει 5 ε, συμβαστικές τροπολογίες και δίνω το λόγο στο μοναδικό Φρανσίσκο Μιγιάν Μον. Θα είμαι σύντομος, Είχα την ευκαιρία να να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία του Φεβρουάριου των δύο αυτών εκθέσεων. Το ένα έχει να κάνει με την συνένεση, εκεί δεν υπήρξαν τροπολογίες και μετά είχαμε τη μη νομοθετική πρωτοβουλία. Όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, εκεί είχαμε 62 τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι από τις 62 αυτές τροπολογίες 14 είναι δικές μου, διότι θέλω να συμπληρώσω κάποια στοιχεία. Ε, είχαμε, περιορι... είχαμε περιορισμένο περιορισμό χώρου, οπότε αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε τροπολογίες γιατί δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε στο αρχικό κείμενο. Οι τροπολογίες που δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με δικές μου πρωτοβουλίες είναι γύρω στις 50. Ε, κάποιες ε, ε, πολιτικές ομάδες δεν έχουν υποβάλει τροπολογίες. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από συγκεκριμένες ομάδες Πέντε συμβαστικές προτάσεις έχω υποβάλει εγώ. Αυτές οι προτάσεις ε, είναι, ήταν αντικείμενο ε, συμβασμού με τους, ε, αυτούς που είχαν υποβάλει τροπολογίες για το πολυπολιτιστικό επίπεδο, το πολυπολιτιστικό επίπεδο ναι, στην Αυστραλία με τον κύριο Τάνο και για τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εμπορική εμπορικών συναλλαγών. Έχω συμφωνία με τον κύριο Καστάλη και Πέτερη. Δεν μπορούσα να συμπεριλάβω την τροπολογία του κύριου Σουέλη. Τώρα για την κυβερνοασφάλεια. Ο κύριος Πάρη, ο κύριος Τάνοκ πάλι οι τροπολογίες του λήφθησαν υπόψη για τα δικαιώματα των ηθαγενών. Και εδώ είχαμε τροπολογίε ε, Ασής, ε, Σολέ και Τάνοκ και δική μου τροπολογία. Και για την κλιματική αλλαγή επίσης έχω οματοποιήσει μια σε τροπολογία του κύριου Πέτερλε και Τάνοκ αυτές οι συμβαστικές ε, τροπολογίες είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού, όπως είπα, με τους, ε, ε τους, τους βουλευτές που έχουν πάλι τροπολογίες, αλλά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς για το επικοινωνικό του πνεύμα, για την ανοιχτή τους διάθεση, για να βρεθούν συμβιβασμοί. Τώρα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που δεν μπαίνουν στο πεδίο των συμβασμών. Θα αναφερθώ σχετικά εν συντομία υπάρχουν και εδώ κάποια μπλοκ, κάποιες τροπολογίες έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία υπήρχαν στις δικές μου τροπολογίες ήδη. Οπότε εγώ προτιμώ τη δική μου διατύπωση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα σας εκπλήξει αυτό. Κάποιες άλλες ε, ουσιαστικά πολύ λίγα πράγματα προσθέτουν, ε, επαναλαμβάνουν κάποια πράγματα. Νομίζω πως δεν είναι απαραίτητες, διότι ουσιαστικά ε, πλήττουν την ισορροπία του κειμένου αναφορά παραπομπή σε συγκεκριμένους οργανισμούς, σε συγκεκριμένα έγγραφα ε, της ε, κυβέρνησης της Αυστραλίας. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στη σχέση με Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αυστραλίας και όχι να μπούμε σε ζητήματα εσωτερικά της Αυστραλίας. Τώρα υπάρχουν άλλες τροπολογίες όπου διαφωνώ. Διαφωνώ κάθετα ε, ζητήματα από των οποίων εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω όχι μόνο επειδή διαφωνώ, αλλά ορισμένε φορές ε, ε, ουσιαστικά καταργούνται δικές μου ιδέες. Ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες δηλαδή που ζητούν να αφαιρεθούν δικά μου επιχειρήματα. Δεν θέλουν να υπάρχει αναφορά στην ευθυγράμμιση της, πολιτική της Αυστραλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των κυρώσεων προ τη Ρωσία. αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είναι κάτι που δείχνει, που αποδεικνύει την προσέγγιση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία σε θέματα εξωτερική πολιτική και νομίζω ότι η έκθεση πραγματικά θα έχανε τη αξία τη εάν ε, δεχόμασταν αυτέ τι τροπολογίε. Υπάρχουν τώρα και άλλε τροπολογίε που και πάλι κατά υπερβολικό τρόπο αναφέρεται στο θέμα, αναφέρεται στο θέμα της μετανάστευσης. Δεν νομίζω να πρέπει να επικεντρωθούμε σε, ε, τόσο πολύ, σε τόσο λεπτομέρειες στο θέμα αυτό, διότι επαναλαμβάνω αυτό πλήττει την ισορροπία του κειμένου και δεν πρόκειται να υποστηρίξω και αυτές τις τροπολογίες. Νομίζω ότι ε, στο αρχικό κείμενο καλύπτονται όλα αυτά και δεν χρειάζεται να ε, το τονίσουμε περισσότερο. Τώρα υπάρχει μια προφορική τροπολογία επικαιροποίηση του κειμένου, διότι 8 Μαρτίου στη Σαντιάκου της Χιλής ε, υπεγράφει η συμφωνία, ε, τη εταιρική σχέση ε, του ειρηνικού, ε, όπου όπως ξέρετε μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ είχε δεχθεί ένα πλήγμα, τελικά όμως η υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Δεν μπόρεσα εγώ όμως να το συμπεριλάβω στο αρχικό μου κείμενο διότι, είναι, διότι εγώ το, το συνέταξα πριν την υπογραφή οπότε υπάρχει αυτή η προφορική τροπολογία που το αναφέρει. Αυτά είχα να σας πω. Αναμένω τα δικά σας σχόλια και αν έχετε ερωτήσεις ευχαριστώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ Φρανσίσκο. Και τώρα οι σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Ασής ε, για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Εκτός μικροφώνου όμως ο κύριος Ασής. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Και δεν ακούμε το κύριο Ασίσο. Ίσως πιο άλλο μικρόφωνο να λειτουργεί καλύτερα. Ναι, μια και έχω την... Να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει μια βασική συμφωνία με την κατεύθυνση ανατολισμού μας και αυτή της, της έκθεσης. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να συζητήσουμε με μεγάλη ε, ε ευχαίρεια και με τον εισηγητή και τον οποίο συγχαίρω για τη δουλειά του. Έχουμε επανειλημμένα μπορέσει να, συζητήσει, να συζητήσουμε ε, τα θέματα και τώρα έχουμε και το τελικό ε, ε, ε σχέδιο που ο, συμφωνεί, ενισχύει τους πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με την Αυστραλία. Υπάρχουν γεωοικονομικοί και γεωπολιτικοί λόγοι σαφείς, γι' αυτό και οι εξελίξεις ε, δικαιολογούν την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία και ο εισηγητής τονίζει όλα όσα συνδέουν αυτές τις δύο περιοχές. Είναι μια μεγάλη περιφέρεια η Αυστραλία ε, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς έχουμε υποβάλει μια τροπολογία όσον αφορά τους, αυ, τους αυτόχθονες ε, λαούς, όπως το, ε, τους αβορήγινες δηλαδή. Είναι περίπλοκο το θέμα και τα τελευταία χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν κάνει θετικά βήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να τονιστεί, να αναφέρουμε το πρόβλημα και να χαιρετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει ε, αντιμετωπιστεί και δεν έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες γιατί στην πράξη αναγνωρίζουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του κειμένου, συμφωνούμε και συμφωνούμε συμφωνούμε και με τις παρατηρήσεις ε, του εισηγητή. Όπως συμφωνούμε και με τα όσα απέρριψε και για τους λόγους στους οποίους τα απέρριψε. Υπάρχει μεγάλη σύντοση απόψεων και άρα θα φανεί αυτό και στην αυρινή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Assis. Ευχαριστώ τον κύριο Ασής. Ο κύριο Τάνοκ έχει τώρα το λόγο. Και ο εισηγητής επίσης. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομο ε, και τηλεγραφικό, θα έλεγα. Θέλω να συγχαρώ τον παλαιό μου φίλο, τον Φρανσίσκο Μιλιαμό, ε, για την ε, έκθεση αυτή. Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά ο συντονιστής είμαστε ικανοποιημένοι ήδη με την αρχική μορφή του κειμένου. Είναι μικρέ οι αλλαγέ που έχουν επέλθει έκτοτε και θετικέ. Ε, έχουν συμπεριληφθεί και κάποιες τροπολογίες μου στους, συμβαστικ... στους συμβασμούς. Είχαμε την υπογραφή ε, της ε, Συμφωνίας του Ειρηνικού που έτσι ανανεώθηκε προς έκπληξη όλων μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ. Ε, οπότε εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ όλων των συμβασμών ε, και θα υποστηρίξουμε γενικότερα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Θέλει κάποιος άλλος ε, τον λόγο. Ο κύριος Αλαφράγκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση του κυρίου Μον. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι όντω αυτή η συμφωνία πλαίσιο θα ενισχύσει σημαντικά τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία. Είναι ένα εταίρο ε, που συμμετέχει σε όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις στο πλάι μας, ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, γίνεται αναφορά στην έκθεση, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, είναι ενεργός ο ρόλος της Αυστραλίας και για τη Συμφωνία των Παρισίων, ο μεταναστευτικός διάλογος με την Αυστραλία, που μια χώρα που έχει μια μεγάλη δυνατότητα υποδοχής και βεβαίως ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις ε, όπου όπως είπε ο κ. Μιγιάν στην έκθεσή του η Αυστραλία συμμετείχε και σε αποστολές διαχείρισης κρίσεων ε, στην ίδια την Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πολύ έτσι, έφορο το πεδίο ε, και για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου αλλά και εν ώψη μιας εμπορικής συμφωνίας όπου πραγματικά εδώ ο εισηγητής προσεγγίσει το θέμα με μεγάλη ευαισθησία, όπως όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπάρχουν, όπως όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπάρχουν ευαίσθητα σημεία και τις δύο πλευρές. Θα ήθελα να ζήσω από τον εισηγητή, εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο, να κάνει κάποιο σχόλιο, να μου δώσει κάποιο στοιχείο ενδεχομένω που θα έχει στη διάθεσή του για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το Brexit την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας. Ε, δεν είναι βεβαίως θεμελιώδες ζήτημα, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια ειδική σχέση με τη χώρα αυτή και δεν ξέρω εάν μπορεί να αξιολογηθεί και αυτό, εφόσον βεβαίως θεωρείται ότι είναι σκόπιμο. Πάντως έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, σοβαρή και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ωραία, δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Να δώσω... Τσάρλς, έχεις και άλλο ερώτημα. Ναι, όχι, για να απαντήσω στον συνάδελφο, τον κύριο Σαλαφράνκα. Δεν ήθελα να μιλήσω για τον Brexit. Ε, το είπα στην αρχή, νομίζω. Ε, βεβαίως, το μεγάλο παράδοξο εδώ είναι ότι αυτοί που είναι υπέρ του σκληρού Brexit στον Βασίλειο επιμένουν ε, ότι ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν ειδική σχέση ε, και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να ξυπνήσουν. Ε, ήρθε εδώ η Πρωθυπουργό τη ε, Αυστραλία, είπε ότι η Αγγλία θα μπει στην ουρά όπω όλοι οι άλλοι για συμφωνία δευτερών συναλλαγών. Ε, και βεβαίω η μεγάλη αγορά είναι η εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 σε ό,τι αφορά την οικονομική ισχύ ε, και το πόσο ενδιαφέρον θα δείξει η Αυστραλία. Ε, η ιδέα δηλαδή ότι η Βασιλεία θα συνεχίσει έτσι το εμπόριο με τις χώρες της πρώην ε, να ανοικοδομήσει το Commonwealth, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εμπορικό μπλοκ, αυτό είναι άλλο ένα από τα ψέματα, άλλη μία ψεύτικη υπόσχεση από αυτούς που υποστήριζαν το Brexit. Ο κύριος Κόξ πήγαινε να τον κόσμο και έλεγε ότι θα έχουμε εκατοντάδες συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών με αυτές τις χώρες ε, του Commonwealth ε, και τώρα έχει σοκαριστεί ε, διότι οι επικεφαλείς των χωρών του Commonwealth θα συνοντηθούν σύντομα και είχε την ιδέα ότι τότε θα, θα προχωρήσει η ιδέα του και του ελέγχθη ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρου των χωρών της Commonwealth ε, να πάρουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως βασικός εμπορικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλη λοιπόν αυτή η ιδέα δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ βεβαίω ε, είμαι πανευτυχή, το λέω εδώ και καιρό. Οι αγγλόφωνε χώρες όπως ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία είναι στην ουρά για να έρθουν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς τον Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώ χωρίς. Φανταστείτε στην Ισπανία να γίνει μια εκστρατεία να φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή με τη Λατινική Αμερική εσείς μπορείτε μόνοι σα να έχετε εμπορική επιτυχία. Αυτό συνέβη με τους ε, οπαδούς του Brexit και τώρα ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε. Ε, και χαίρομαι που συμβαίνει αυτό, γιατί το λέω και χρόνια είναι ε, μόνο στα μυαλό του, του Ντάνιελ Χάνον αυτά τα περί Commonwealth. Ευχαριστώ. Ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή Ο Κύριε Μικιάν Ευχαριστώ Πρόεδρε και σύντομα. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ και με τη σειρά στον κύριο Ασής, σας σκιώδη από τους σοσιαλιστές. Ε, χαίρομαι για τις ε, επαφές και τη συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και για τα δικαιώματα των ε, αβοριγένων βρίσκουμε μια κοινή γλώσσα επιτέλους και από το 2008 έχουμε αναφερθεί ε, σε αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Αυστραλίας για ε, την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και υπερβολικά και με τον συνάδελφο Τσάστα που είμαστε εδώ παλιά από το 2004, γι' αυτό είναι υπερβολικό στους επένους τους και διθυραμβικός ε, σε ό,τι με αφορά. Πολλές από τις τροπολογίες του τις έχω συμπεριλάβει στο συμβασμό. Ο Τσάλις έχει κάνει περισσότερες τροπολογίες και από τους πρώτους, γι' αυτό φυσικά έχω συμπεριλάβει. Σε ό,τι αφορά τον Νάτσο Σαλαφράνκα, θέλω να τον ευχαριστήσω δεν μας εκπλήσει, δεν εκπλήσει κανένα ότι συμφωνούμε και ε, στην ουσία και στον τύπο γιατί είμαστε κοντά ε, όχι μόνο λόγω χώρας αλλά και πολιτικής παράταξης κλπ. Σας ευχαριστώ όλους. Χαίρομαι που συμπίπτουμε επί της ουσίας. Αυτό τώρα το θέμα για το Brexit. Απάντησε εξ ονόματος μου κάπως ο Τσαρ Στάνοκ. Κοιτάξτε, ειλικρινά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι οι σχέσεις Αυστραλίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασε κατά πολύ τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, που στο παρελθόν ήταν σημαντική βεβαίω λόγω των ειδικών δεσμών, αλλά τώρα είναι σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αυστραλία, όχι με του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτή η συμφωνία πλαίσιο θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως και η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, που θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τους επόμενους μήνες, ελπίζω για να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο, να ευαφηθεί αυτή η σχέση. Θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά Είμαι πεπισμένος ότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει και από πλευρά Αυστραλίας και από εμά. Θα μας λείψουν οι Βρετανοί. Ε, είπα και εγώ, όπω και άλλοι, δεν θέλαμε αυτό το Brexit, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε ε, την απόφαση του λαού. Σίγουρα θα τους λείψουμε κι εμείς. Αλλά οι σχέσεις βρυξελλων Βρυξελών θα παραμείνουν και προσπαθούμε με αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, τη συμφωνία ευθύνων συναλλαγών, να τι εμβαθύνουμε, να συσφίξουμε του δεσμού. Πέρσι άρχισε ε, ένα σχήμα ε, συνεδριάση ηγετών. Εντάξει, θα αφήσει κάποιο κενό το Ηνωμένο Βασίλειο. Φεύγοντα, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω αύριο η ψηφοφορία να ε, καταλήξει σε ένα ισόρροπο κείμενο που να σημειώνει τη σημασία των ε, σημερινών και μελλοντικών σχέσεων ε, Αυστραλίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Φρανσέσκο Μιγιανμόν, για τα καταληκτικά σου σχόλια. Όσο μιλούσε, ζήτησε το λόγο ο κύριος Καστάλντο. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να πεις κάτι μετά ε, τα καταληκτικά σχόλια, αλλά είσαι και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Τι να πω εγώ, φτωχός βουλευτής. Δεν, πειράζει, δεν ζήτησα το λόγο πριν, γιατί επειδή ήμουν σκιώδης, νόμιζα ότι θα μου δίνατε το λόγο σε όλους τους σκιώδης, αλλά δεν πειράζει. Δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ είμαι σε επαφή με τον εισηγητή, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα για τη δουλειά της Επιτροπής. Κύριε Καστάλντο, αν ήσασταν εδώ εκείνη τη στιγμή θα σας είχα δώσει το λόγο. Νομίζω πως ήρθατε ενώ συζητούσαμε, βεβαίω είστε σκιώδη και είστε στον κατάλογό μου, αλλά αν δεν ήσασταν εδώ δεν μπορούσα. Ναι, έφτασα όταν μιλούσε ο κύριος Αλαφράγκα. Στη διάρκεια της Α, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται τώρα να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Έφτασα στη διάρκεια της συζήτηση, δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα, δεν είναι θέμα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει αύριο το πρωί. Στις 20 Μαρτίου. Πολύ ωραία. Πάμε ένα σημείο για σήμερα. Δεν υπάρχει, οπότε τελειώσαμε. Καλό σας απόγευμα. Να ευχαριστήσω τους συναδελφούς που έκατσαν μέχρι τέλους.